για συνομιλίες για το θέμα του Ιράν. Ο Στέφαν Φούλερο, συνάδελφος και φίλος, θα συμμετάσχει στο επόμενο τμήμα της συζητήσεως. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Γκόμες, Συμφωνία Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβύης. Το λόγο έχει για τέσσερα λεπτά η εισηγήτρια η κυρία Γκόμες. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Λιβύα έχει μια στρατηγική θέση όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Πέρα από το ενεργειακό απόθεμα το οποίο έχει που είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάποια κράτη-μέλη έχουν έντονες σχέσεις, βαθιές σχέσεις με τη Λιβύη και έτσι ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γι' αυτό υποστηρίζουμε μια συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις με τη Λιβύη που θα συμπεριλαμβάνει διάφορες δράσεις και διάφορα πεδία από πλευράς πολιτικών. Όμως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η Λιβύη κυβερνάται από ένα δικτατορικό καθεστώς με σοβαρότατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πλήγματα τρομοκρατία σε άλλες χώρες. Και θα πρέπει να βρεθεί η σωστή οδός. Γι' αυτό η συμφωνία πλαίσιο με τη Λιβύη θα μπορεί να εγκριθεί από την Ευρωβουλή μόνο αν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις θα είναι σεβαστοί και σεβαστές ο όρος εκ των όνου να επιτρέψει να ξανανοίξει η ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες στην Λιβύη και με διευρυμένη εντολή. Τολμώ να το πω αυτό με σαφήνεια και κάθετα. Αν δεν γίνει αυτό δεν θα μπορέσει να υπάρξει συμφωνία. Θα πρέπει επίση ε, να κυρωθεί η σύμβαση της, ε, των Ηνωμένων Εθνών της ε, Γενέβη για του μετανάστες. Δεν είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζεται το καθεστώ των προσφύγων από πλευρά τη Λιβύη. Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Λιβύη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη εκείνου που ετούνται άσυλο και χρειάζονται διεθνή προστασία. Και θα πρέπει να εφαρμόζονται όλε αυτέ οι αρχέ με την αρχή τη non-refoulement, τη μη απέλαση. Καθώ επίση επίσης και για τους υπήκους ε, της ε, Ερυθρέας ε, που βρισκόντουσαν στη Λιβύη και τέτοιου είδους γεγονότα δεν πρέπει να επαναληφθούν. Θα πρέπει επίσης με τον καλύτερο τρόπο να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ζωής των δύο εκατομμυρίων μεταναστών που ζουν στην Λιβύη. Πρέπει να τύχουν νόμιμης προστασίας και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως δούλοι, ως σκλάβοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει σε προγράμματα για να αντιμετωπιστεί το εμπόριο ανθρώπων και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών θα πρέπει να ε, ζητηθεί από τις ε, οργανώσεις που εργάζονται με τους μετανάστες ε, στη Λιβύη να βελτιωθούν οι συνθήκες των μεταναστών και να πάψουν να υπάρχουν οι καταχρήσεις που συνέβησαν στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να, να αγνοήσει το θέμα της θανατικής ποινής και θα πρέπει να δημοσιευθεί, να γνωρίζουμε την, το όνομα των υπηκών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει η Λιβύη να κυρώσει το καθεστώς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης. Θα πρέπει να ενθαρρύνει τρόπους και μορφές ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δώσουν τη δυνατότητα στην Λιβύη να δημιουργήσουν μια κοινωνία ελεύθερη και που θα δώσουν τη δυνατότητα θεσμικών δυνατοτήτων για τις ε, ε, ενώσεις επιχειρηματιών, πολιτών κτλ δεν είναι δυνατόν να, πούμε ότι η, σε σχέση με το καθεστώς γκαδάφι θα πρέπει να αντιληφθεί οπωσδήποτε αυτή την ανάγκη που υπάρχει. Επίσης όσον αφορά τον τομέα της υγείας με την Μπενγάζη και με άλλα κέντρα ιατρικής περίθαλψης θα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Έχουμε ε, ε, ε, πληροφορηθεί ότι υπάρχουν εδώ δυσκολίες όσον αφορά την ενεργειακή συνεργασία. Παρ' όλα αυτά θα ήταν ε, θετικό να υπάρξει μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα, ε, ε, θα λειτουργήσει στην Τρίπολη για να συνοδεύσει αυτές τις διαπραγματεύσεις και να υποστηρίξει αυτή την ανάπτυξη των σχέσεων με τη Λιβύη. Ζητήσαμε κύριε Επιτροπέ από την Λιβύη να έχουμε τα αναγκαία στοιχεία για αυτή την συνεργασία με τη Λιβύη. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να διατεθούν αυτά τα στοιχεία σύντομα. Και σε σχέση με την ευκαιρία για την εντολή του Συμβουλίου δεν δυνατόν να παρακάμπτεται το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στο τέλο ε, για τη συνεργασία όλων των σκιωδών εισηγητών, που η συνεργασία του ήταν σημαντική για την εκπόνηση αυτή τη έκθεση, ε, που είναι τόσο δύσκολο. Σα ευχαριστώ. Εξ ονόματος Επιτροπής, ο Επίτροπος ο κύριος ε, Φούλε. Oh, uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώσω το σώμα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ενώσεως Λιβύης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη συνεργάζονται στενά όσον αφορά το θέμα της Λιβύης. Έχουμε κοινό συμφέρον να εξασφαλίσουμε θετικές εξελίξεις όσον αφορά σχέσεις μας με τη Λιβύη που είναι σημαντικός γειτονάς μας. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να συγχαρώ την αντιπροσωπεία σας για τις σχέσεις με το Μαγκρέμπ και ιδιαίτερα για τη συμφωνία που επετεύχθη κατά τη διάρκεια της επισκέψεως στην Τρίπολη που προβλέπει τακτικές διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο της Λιβύης. Είμαι αποφασισμένος να εξασφαλίσω ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμών μας θα συνεχιστεί. Κυρίως θέλω να ενημερώνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τακτικά για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Πλαίσιο. Γνωρίζω ότι ο βασικό μα διαπραγματεύτη ο επικεφαλής διαπραγματεύσεων, σα ενημερώνει μετά από κάθε κύκλο διαπραγματεύσεων, κάθε συνεδρία διαπραγμάτευση, να σα ενημερώσω ε, ποια είναι η πιο πρόσφατη κατάσταση. Ολοκληρώθηκε ο ένατο γύρο διαπραγματεύσεων μέσα Νοεμβρίου στην Τρίπολη. επόμενο γύρος θα είναι 24 με 26 Ιανουαρίου στι Βρυξέλλες από την εκείνη των διαπραγματεύσεων πάνω από δύο χρόνια πριν. Έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο. Έχουμε προσωρινά συμφωνήσει όσον αφορά το προήμιο και έξι από τα δέκα κεφάλαια της συμφωνίας. Πιο συγκεκριμένα, φτάσαμε σε προσωρινή συμφωνία όσον αφορά το κεφάλαιο για τον πολιτικό διάλογο που εμπεριέχει σημαντικές αναφορές στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καταπολέμηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, της καταπολέμηση της τρομοκρατίας κλπ. Πρέπει να σας πω ότι η Λιβύη έχει δεχθεί να υπάρχει τακτικός διάλογος αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που ήταν θεμελιώδης στόχος μας. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι είμαστε άκρος ικανοποιημένοι με το, ε, το αποτέλεσμα αυτό, για το κεφάλαιο αυτό, όπως τα γνωρίζετε υπάρχουν κάποια εκκρεμή ζητήματα όπως το θέμα της ενέργειας και το εμπόριο. Η ενέργεια είναι ο πυρήνας της οικονομίας της Λιβύης, το 70% του ΑΕΠ της χώρας. Οπότε με προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό η Λιβύη και αυτό είναι κατανοητό όσον αφορά το εμπόριο. Έχει περιορισμένη εμπειρία η Λιβύη όσον αφορά την διαπραγμάτευση για περίπλοκες εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό ήταν μέτρια η πρόοδος όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα και οι ειδικοί και τι τις δύο πλευρές συναντώνται τακτικά, πολύ τακτικά για να καταλήξουμε σε συμφωνία επ' αυτών των δύο θεμάτων το ταχύτερο δυνατόν. Υπάρχουν βεβαίως δύσκολα πολιτικά ζητήματα, ένα από αυτά είναι το θέμα του καθεστώτος των τζιγκάνων. Αρνείται κατηγορηματικά η Λιβύη να κάνει ρητή αναφορά όσον αφορά το καθεστώς των τζιγκάνων. Είναι έτοιμη να δεσμευτεί όμως όσον αφορά συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της ατιμορρησίας κυρίως για τα εγκλήματα αυτά που καθορίζονται. Για, το, για τη σύμβαση της Ρώμης, συνθήκη της Ρώμης και για τη μετανάστευση. Ε, σημείωσα τα όσα συνέστησε το Κοινοβούλιο για τη συγκεκριμένη πτυχή των διαπραγματεύσεων και σίγουρα θα το συζητήσω αυτό το θέμα με τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τη μετανάστευση, σας διαβεβαιώ ότι έχουμε δεσμευθεί να εξασφαλίσουμε το ότι η Λιβύη θα σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις σχετικά με την αρχή του νοεφουλμό της μη επαναπρόθεσης. Αυτό είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε επίσης ότι είναι σημαντικό να, το ταχύτερο δυνατόν η Λιβύη να προσχωρήσει στην Σύμβαση της Γενέβης του 1951 και το πρωτόκολλο του 1967 όσον αφορά το καθεστώς των ε, προσφύγων. Όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Λιβύη ανέφερε ότι δεν προτίθεται να προσχωρήσει σε αυτή την σύμβαση. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι ακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ε, της Λιβύης και της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ούτως ώστε να βρεθεί σωστή λύση και αυτός ο φορέας να μπορεί να εκτελέσει πλήρως την αποστολή του ε, σε ασφαλές περιβάλλον. Γενικότερα τον Οκτώβριο καταλήξαμε σε κάποια συμφωνία για να αυξήσουμε τη συνεργασία με τη Λιβύη όσον αφορά όλα τα θέματα που άπτονται της μεταναστεύσεως συμπεριλαμβανομένης και της διεθνούς προστασίας βελτιώνοντας τις συνθήκες για τους μετανάστες στη Λιβύη τη διαχείριση των ε, μεταναστών και του ελέγχου των συνόρων. Είναι θετική εξέλιξη διότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τη Λιβύη για να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σχετικά με τη μετανάστευση. Τέλος, κύριε Πρόεδρε και εξότιμα μέλη, θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, εντολές διαπραγματευτικές που ζήτησε το σώμα, το μνημόνιο ε, λοιπόν, το άρθρο 218 της Συνθήκης της Λισαβόνας ε, προβλέπει κάτι τέτοιο και αυτός, ε, αυτό το μνημόνιο κατανόησης είναι κάτι που έχει ζητήσει το Συμβούλιο και έπρεπε να μελετήσει το έτοιμά σας σε οριζόντιο επίπεδο θα ήθελα να σας πω με τα χαράς ότι αυτή η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί και όπως πιθανότατα θα γνωρίζετε το Συμβούλιο έχει δώσει πρόσβαση όσον αφορά αυτές, αυτό το μνημόνιο κατανόηση για τη σύναψη τη συμφωνία με τη Λιβύη, σεβόμενοι πάντα ε, τους κανονισμούς περί ασφαλείας του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο έχει ενημερώσει τον Πρόεδρο ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων δεόντως. Αυτά και ευχαριστώ για την προσοχή σα. Εκ των πολιτικών ομάδων, ε, για το Λαϊκό Κόμμα, ο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. The Council of June 2009 το Συμβούλιο του 2009 συνέστησε κάποιε προτεραιότητε, δηλαδή τη σύναψη συμφωνιών επανεισδοχή με τη Λιβύη και την Τουρκία. Και θεωρήθηκε ότι πρόκειται για πύλες, σημεία εισόδου μίζωνα. Η δε πύλη της Λιβύης ε, έχει σχέση με Μάλτα και Ιταλία. Όμως απειλείται να αλλοιωθεί η δημογραφία της Μάλτας. Έχει αναγνωριστεί το ότι θεωρητικά όλοι έχουμε συνυπευθυνότητα, όμω στην πράξη τίποτα δεν γίνεται για να διορθωθεί η κατάσταση. Ο αριθμό των αφήξεων στη Μάλτα μειώθηκε μόνο όταν η Ιταλία που και αυτή πλήσεται συνήψε διμερή συμφωνία με τη Λιβύη. Και η Λιβύη ανέλαβε να περιπολεί τα χωρικά τη. Και έχουμε λοιπόν μια συμφωνία πλαίσιο και μια συμφωνία πανεσδοχή. Οι διαπραγματεύσει τώρα που προχωρούν είναι δύσκολε, αλλά εμεί στηρίζουμε τι προάθειε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίση ενθαρρύνουμε την συνέχιση ε, ω την τελική επιτυχία. Και εμεί έχουμε προτείνει να συνηθεί ε, μεταναστευτική συμφωνία τον Οκτώβριο για μα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Έτσι θα προετοιμαστεί η χώρα για κάποια ζητήματα όπω ένα σύστημα προστασία για, για το άσυλο. Ε, νομοθεσία σε σχέση με την Αφρικανική Σύμβαση για πρόσφυγες και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Γνωρίζουμε την κατάσταση των αρμενικών δικαιωμάτων, ξέρουμε δεν υπάρχει αναισθησία του τύπου, ξέρουμε ότι υπάρχει κακή μεταχείριση κρατουμένων, βασανιστήρια και θανατική ποινή. Όμως η επανεισδοχή χρειάζεται. Αυτό βέβαια εξαιρεί όσους θέλουν πολιτική προστασία, δικαιούνται άσυλο, κινδυνεύουν να ε, υποστούν ε, απειλή υγείας θανάτου στην, στη χώρα, αλλά κατά τα άλλα ισχύει η αρχή της επαναπρόθεσης, ο κ. Παντσέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η δουλειά που έκανε η Άννα Γκόμες είναι σοβαρή συνεισφορά σε αυτά πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό της Συμφωνίας Πλαισίου διαδραματίζει η Λιβύη αναφεσβήτητα αποφασιστικό ρόλο στην καταπολέμηση τη Τρομοκρατία, την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αφρική, την καταπολέμηση τη παράνομης μετανάστευση στη Μεσόγειο και στον ενεργειακό τομέα. Γι' αυτό στόχο μα στα πλαίσια τη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα πρέπει να είναι να παγιώσουμε την ένταξη τη Λιβύη σε πολιτικό και οικονομικό σύστημα διεθνέ που θα βασίζεται σε κοινού κανόνε. Για να πραγματοποιήσουμε αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που θα επιβληθούν στη Λιβύη και παίρνει συστάσει. Και όσον αφορά το θέμα τη μετανάστευση, η Λιβύη σήμερα αντικειμενικά πρέπει να πούμε είναι χώρα διέλευση. Είναι θέμα πολύ σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε μόνο από το θέμα από την πλευρά τη ασφάλεια ε, δηλαδή επαναπροωθήσεις και σταμάτημα μας μετανάστευσης. Χρειάζεται μια κυβέρνηση που μπορεί να, ε, να έχει οικονομική κατάσταση, κοινωνική κατάσταση που να μπορεί να, κάπως να σταματήσει αυτή τη ροή και θα πρέπει η Λιβύη να, να υπογράψει τη Σύμβαση τη Γενέβη και υπάρχει και το πρόβλημα τη πανεισδοχή των μεταναστών. Βάσει εγγύσεων για την ασφάλειά του όσον αφορά τι συνθήκε διαβίωση των ε, μεταναστών. Μετά είναι και το θέμα τη μεταρρύθμιση οικονομική και τη δημοκρατική που θα επιτρέψει σε αυτή τη σημαντική χώρα να ε, διευρύνει τον, περισσότερο το δημοκρατικό τη χώρο. Και αυτό να το λάβουμε υπόψη όλο και περισσότερο όπω αναφέρει, το είδαμε να συμβαίνει και στη γειτονική την Και τέλο αυτή η σύσταση μα οδηγεί στο να σκεφτούμε τι γίνεται με τι επαφέ και συμφωνίε. Αυτέ συμφωνίε μπορούν να δώσουν ε, μια συνεισφορά για να επιληθούν τα προβλήματα όμως δεν ε, λύνουν μόνο σε αυτές τις συστάσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχουμε με τα λιευτικά σκάφη ιταλικά δείχνει ότι, το οι διμερεί συμφωνίες αφήνουν εκρεμή κάποια προβλήματα. Μετά τίθεται και στα τα πλαίσια της αναθεωρήσεως της πολιτικής γειτονίας και θα πρέπει να εξετάσουμε ένα νέο πλαίσιο για τη Λιβύη. Θα πρέπει λοιπόν να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις και στον πληματισμό το Κοινοβούλιο έχει δώσει εντολή το Συμβούλιο όσον αφορά τη διαμόρφωση πλαίσιο και σε αυτή τη φάση θα πρέπει λοιπόν αγαπητέ Επίτροπε, να αλλάξει ο ρυθμός και θα πρέπει και να συμμετέχει όλο και περισσότερο το Κοινοβούλιο στη διαμόρφωση νέων πολιτικών που στρέφονται προς τον νότο της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Η κυρία Οζουλάντ, ε, εκ μέρους των Φιλελευθέρων, για 1,5 λεπτό. Thank you. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα, να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για την εξαιρετικό του έργο το οποίο επετέλεσε και έτσι αποξαλώθηκαν οι θέσει όλων των ομάδων του Πολιτικού Κοινοβουλίου. Σε αυτή την έκθεση θέλω να σα τονίσω το πόσο σημαντικό είναι να συζητήσουμε το τι κατάσταση περνά, τι κατάσταση διέπει του μετανάστες τη Λιβύη όταν έρχονται στην Ευρώπη, προσπαθούν να διασχίσουν την Μεσόγειο και καταλαβαίνω το ότι και οι νότιες χώρες ε, ανησυχούν όσον αφορά αυτές τις μεταναστικές ροές γιατί και αυτό είναι πίεση στον προπολογισμό του και την κοινωνία του. Όμω θα πρέπει να μην ξεχνούμε τα συμφέροντα των κρατών μελών, ε, χωρί να παραβλέπουμε και τι ευρωπαϊκέ αξίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντέχει να βάψει τα χέρια της κόκκινα με το αίμα των, ε, του Ντοράσιλο και των λαθρομεταναστών. Επομένως, δεν θα πρέπει καμία συμφωνία να δείξει σε απάνθρωπη συμπεριφορά, σε βασανιστήρια, σε εκτέλεση και για αυτό με μεγάλη μου χαρά άκουσα από εσάς, Επίτροπε, ότι βλέπετε να υπάρχει μια πρόοδο στις σχέσεις με τη Λιβύη. Ευχαριστώ. Είδαμε στην Τινησία τι έγινε. Εξεγέρθηκε ο λαός κατά του καθεστώτος του καταπιεστικού που του στέρισε τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα επί χρόνια είναι πηγή ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί επί σειρά ετών υποστηρίζαμε αυτή τη δικτατορία. Για να χειροτερέψουμε τα πράγματα, μπορεί να διαπράξει το ίδιο πρόβλημα και στη γειτονική χώρα τη Τινησία, τη Λιβύη. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο αλλάξουν πορεία, θα εξακολουθούν να υποστηρίζουν άλλον ένα δικτάτορα στην περιοχή εν ονόμα τη αθερότητα και του ελέγχου των συνόρων και τη μετανάστευση. Ψηρά ετών το καθεστώ του πηγείται ο Καντάφη, ένα του καλύτερου φίλου του Μπενάλη, όπω είδαμε και τώρα, συστηματικά παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών του και κυρίω των μεταναστών εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά, τα Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια κράτη είχαν στενότερε σχέσει με την Λιβύη και τώρα διαπραγματευόμαστε αυτή τη συμφωνία πλαίσιο. Γι' αυτό παροτείνω το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, σημειώσουν, να δουν τι μελη γεννάστε και θα πρέπει να τεθούν κάποιε προποθέσει πριν τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνία με τη Λιβύη. Η Λιβύη θα πρέπει να επικυρώσει και να εφαρμόσει την συμφωνία, τη σύμβαση ε, τη ΥΠΑ τη Αρμοστία του ΟΗΕ για του πρόσφυγε και να επιτραπεί στο φορέα να μπει στη χώρα. Θα πρέπει να προστατεύονται οι μετανάστε και θα πρέπει να υιοθετηθεί νομοθεσία για, την, ε, για του άσυλο και αρχή του νόμου Δεν μπορεί να υπογραφεί καμία συμφωνία μέσω του να μην καταργηθεί η κατάσταση επικρατεία του που υπόκειται σε απάνθρωπη μεταχείριση. Και αυτό θα αργήσει να γίνει, πιστεύω, και αυτό θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, μην προωθήσει τη συμφωνία την επανιστοχή. Θα πρέπει και το Κοινοβούλιο στι διαπραγματεύσει συμμετέχει πλήρω. Οι πράσινοι έχουν ισχυρέ ε, αντιρρήσεων αφορά συμφωνία ε, μυστική με τον Καντάφη πίσω εις βάρος των μεταναστών. Κάτι τέτοιο δεν αποκρίνεται στι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ενώσης ούτε στι ούτε εξυπηρετεί τα μακρότερα συμφέροντά τη στην περιοχή. Το είδαμε τι έγινε στην Τινησία. Μόνο δημοκρατική και ελεύθερη χώρα θα είναι πραγματικά σταθερή και πλούσια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να κάνει δύο φορέ το ίδιο λάθο. Ευχαριστώ. Εκ ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε είναι μια χώρα Λιβύη όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται ως ε, ε, ε, συνήθεια καθημερινά και πραγματικά τα πολιτικά κόμματα έχουν απαγορευτεί. Ο Καδάφη είναι ο Φιντέρ Κάστρο της Αφρικής προσπαθεί να δώσει την εικόνα ενός ε, καλού πατέρα που ε, προσέχει για τα παιδιά του. Εμείς όμως ε, στη χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρουμε ότι συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Είναι ένας υποστηρικτής των τρομοκρατών, όπως αποδείχθηκε και με το, τη βομβιστική απόπειρα στο αεροπλάνο της Παναμ που έπεσε στο Λόκεμπι. Και πρέπει εδώ να διασφαλιστεί ότι θα βρίσκεται εκτός της προσπάθειας σε σχέση με τα, τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρει ε, πρόσβαση στα πετρελαϊκά αποθέματα της Λιβύης. Ωστόσο, λόγω πραγματιστικών αναγκών δέχομαι την ανάγκη να υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις ε, με τη Λιβύη υπό μια συμφωνία πλαίσιο. Όμως αισθάνομαι ότι όλα όσα κάνουμε είναι παγιώνουμε την εξουσία του Γκαντάφη που όταν θα έρθει η ώρα θα δώσει την εξουσία σε έναν από τους ε, γιους του ώστε να συνεχιστεί αυτή η σταδιοδρομία. Κύριος Χατζηγεωργίου να ευχαριστήσω αρχικά την ε, δουλειά που έγινε από την εισηγήτρια. Να ευχαριστήσω για την παρουσία του κυρίου Φούλε εδώ. Θεωρούμε πως στην ευαίσθητη από κάθε άποψη περιοχή της Μεσογείου θα πρέπει να γίνονται συνεχείς προσπάθειες για ανάπτυξη της κατανόησης και της συνεργασίας. Μια συνεργασία σε ισότιμη βάση που να λαμβάνει υπόψη τις ασυμμετρίες και ανισομέρειες που υφίστανται στου διάφορου τομεί ανάπτυξη ανάμεσα στι χώρε τη μεσογείου και ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ένωση και τι γειτονιάζουσες σε αυτή χώρε τη περιοχή, Μια συνεργασία που να στενοχεύει στην επικράτηση τη Ειρηνή. αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάλογο στη βάση του αλληλοσεβασμού και πρέπει ω εκ τούτου να είμαστε ανοιχτοί στην αλληλεπίδραση. σε αυτό το πλαίσιο είμαστε υπέρ ενδυνάμωσης των σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη λιβύη υπάρχουν ωστόσο ορισμένα ευαίσθητα θέματα τα οποία πρέπει να προσεχτούν ιδιαίτερα στη διαδικασία ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. θα σταθώ κυρίω στο θέμα των προσφύγων των μεταναστών και τη συμφωνία επανεισδοχή. επιδιώκεται να υπάρξει συμφωνία επανεισδοχή με τη λιβύη ω μέρο τη συμφωνία πλαίσιο που συζητείται μεταξύ ευρωπαϊκή ένωση και λιβύη. μια ενδεχόμενη υπογραφή μια τέτοια συμφωνία χωρί παράλληλα να υπάρξουν μεταρρυθμίσει που να βελτιώνουν την κοινωνικο οικονομική πραγματικότητα των μεταναστών θα προσθέσει στη συνέχιση της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και θα συνηγορήσουμε έτσι στην εξαναγκαστική επιστροφή των μεταναστών σε συνθήκες που δεν εγγυούνται την ασφάλειά τους ούτε διασφαλίζουν τα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα διαβίωσης. θα πρέπει να ζητηθεί από τις λιβικές αρχές όπως αναγνωρίσουν νομίμως την παρουσία της ΥΠΑ της αρμοστίας του οηε για τους πρόσφυγες και θα πρέπει επίση να σταθούμε στο ευαίσθητο θέμα τη θανατική ποινή θα ήταν ορθό να επιδιωχθεί συμφωνία αναστολή τη εφαρμογή τη στη λιβύη με απότερο σκοπό την κατάργησή τη. ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι υπέρ τη συνάψεω συμφωνία πλαισίου μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Λιβύη, διότι αντιπροσωπεύει μία πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν επί σημείων όπως η μετανάστευση, η συνεργασία οικονομική και υγειονομική, κυρίως στην καταπολέμηση του AIDS και εν μέρη όσον αφορά το ενεργειακό πρόγραμμα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ο έλεγχο που ασκεί η Λιβύη όσον αφορά τι τρομοκρατικέ δραστηριότητε, όχι μόνο εντό τη ίδια επικράτειά τη, αλλά και επί των νοτίων συνόρων τη χώρα ε, στα βόρεια σύνορα τη χωρα Έγινε συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και τη κυβερνησεω τη Λιβύη επί των γενικών αρχών οπω είναι το τον Ρώμα και το καθεστώς των προσφύγων. Πορά παραμείνουν να γίνουν, αυτό είναι προφανές, αλλά είναι σημαντικό να υποστηρίζει την συμφωνία που ήδη έχει διαπραγματευτεί χωρίς να την αφισβητήσει γιατί αλλιώς διακινδυνεύουμε να χάσουμε τα επιτευθέντα αποτελέσματα. Εύχομαι στη συνεργασία μεταξύ Λιβύης και Ευρωπαϊκής Ενώσεως να πετύχει τα ίδια αποτελέσματα όπως και απέρευσαν και τη συμφωνία φιλίας μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης που ε, έκλεισε και γύρισε σελίδα όσον αφορά το απεικιοκρατικό παρελθόν. Λοιπόν, θα πρέπει να εξεταστούν συγκεκριμένα θέματα, ε, πρέπει να μπορούμε να επιλέξουμε τους συνομιλητές μας. Ε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό το κράτος εγκληματία και με τον Γκαντάφη έχει μεριμνήσει για την εξαγωγή ε, προϊόντων. Δηλαδή κερδίζει όχι μόνο από το πετρέλαιο αλλά και εκβιάζοντας την Ευρώπη. Ο δικτάτορας ε, Γκαντάφη πήρε εκατομμύρια εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται η προσπάθεια να τον λαδώσουμε για να μην έρχονται πρόσφυγες, μετανάστες και πρόσφυγες στην Ευρώπη. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει αυτό να το λάβει υπόψη ε, και να μην ε, εμπιστεύεται τόσο πολύ τον Καντάφη. Εγώ δεν τον εμπιστεύομαι. Τέσσερα δισεκατομμύρια έχει πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι ο Καντάφη όλο και περισσότερα χρήματα θέλει να πάρει ώστε να αποφευθεί να γίνει μια μαύρη ήπειρος η Ευρώπη να κατακλειστεί από, από μετανάστες. Θα πρέπει εδώ να δούμε ότι όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί έχει ε, παρακολεί εκατομμύρια ε, ε, Αφρικανούς να προσθέθουν, να μεταφούν στην Ευρώπη και γι' αυτό εισπράττει τεράστια ποσά. Δεν θα πρέπει όμως να ανταμείβεται ο Γαδάφη αλλά να τιμωρηθεί διότι αφήνει αυτές, αυτούς τους ανθρώπους ανεξέλεγκτα να προσέρχονται στην Ευρώπη και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να επιστρέφουν στην χώρα αυτή οι όσοι ήρθαν από εκεί. Πρέπει πολλά περισσότερα να γίνουν και αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτών που προσπαθούν να περάσουν τη Μεσόγειο και να καταλήξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχει πραγματικά ασκεί την δύναμη του μαγνήτη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους ανθρώπους. Ε, πρώτος είναι ο κύριος Σβένσον για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Λίμπια τα πάει πάρα πολύ αφορά την κύρωση των διεθνών συμφωνιών. Όμω ε, επίση έχουν καλέ επιδόσει στην μία εφαρμογή του και είναι ένα σκάνδαλο το ότι έχουν μέλο στο Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα Ανθρωπίνα Δικαιώματα το ίδιο για τη Σαουδική Αραβία. Είναι σημαντική μα εμπορική εταιρεία, άρα θα πρέπει να του αναγκάσουμε να φροντίσει περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι βασικέ θεμελιώδει ελευθερίε θα πρέπει επομένως να συζητήσουμε και για τους πρόσφυγες και πώς τους ε, μεταχειρίζονται. Συμβούλιο, Κομισιόν δεν μπορούν να, να αναπείσουν τη χώρα, ε, να δεχθούν εκπροσώπους της ΥΠΑ της ε, Θα συνεχίσει η κατάσταση. Μια που ξέρουν πάρα πολλά την τέχνη του να ξεγελάνε, είναι αναξιόπιστη. Και τι θα γίνει με αυτή την συμφωνία πλαίσιο. Τι πάει να πει πλαίσιο όσον αφορά το μυαλό των ε, ανθρώπων του καθεστώτος. Ούτε όρια ξέρουν, ούτε κανένα πλαίσιο τους ρυθμίζει και τους συγκρατεί γιατί ε, δυσμενείς διακρίσεις, βασανιστήρια, ε, ρατσισμός κατά των ε, Αφρικανών όλα αυτά σοβούν στη χώρα. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι ανθρώπινες ελευθερίες και τα δικαιώματα να τους απειλήσουμε, να τους πιέσουμε ούτως ώστε οι απάνθρωπες συμπεριφορές να σταματήσουν. Γιατί αυτό το επιβάλλει η συνθήκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε. Η Λιβύη είναι ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος ε, φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μίζων εμπορικό εταίρος. Περισσότερο από δύο τρίτα του όγκου των εμπορικών συναλλαγών της Λιβύης ε, πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατάφεραν οι αρχές αυτής της χώρας να πάυσουν το καθεστώς απομόνωσης στο οποίο είχαν βρεθεί. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για οικονομικά συμφέροντα. Πρόκειται και για αξίε και αρχέ που δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε λόγω μια πραγματιστική ή ρεαλιστική προσέγγιση. Η Λιβύη δεν υποστηρίζει πια τα ατομικά όπλα, τα πυρηνικά όπλα ή τους ε, τρομοκράτες και οι ε, βούλγαρες νοσοκόμες απελευθερώθηκαν και όσον αφορά τις κατηγορίες για μόλυνση πολιτών ε, με AIDS από αυτές, αυτό έχει εγκαταληφθεί. Πρέπει τώρα να δούμε για αυτές τις σχέσεις με την Λιβύη χρειάζεται ένα ηθικό πλαίσιο το οποίο θα είναι βιώσιμο. Η έκθεση της κυρίας Γκόμες καταδεικνύει πόσο σημαντικές είναι οι ελλείψεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να καταπολεμηθεί αυτή την, η κατάσταση. Πέρσι εγκρίναμε ένα ψήφισμα που ζητείται από τη Λιβύη να πάψει να ασκεί την θανατική ποινή, να επιβάλλει τη θανατική ποινή. Πρέπει να εμείνουμε και να επιμείνουμε και να απαιτήσουμε να συμμορφωθεί η Λιβύη με, ε, με το διεθνές αυτό καθεστώς των αρχών που πρέπει να σέβεται. Και το πρόβλημα των μεταναστών και των ε, προσφύγων είναι πάρα πολύ σημαντικό επιστρέφουν αναγκαστικά στις χώρες προέλευσής τους και εκεί ε, υπάρχει πραγματικά ελοχεύει σημαντικότατος κίνδυνος για αυτούς. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση λοιπόν η Λιβύη να εγκρίνει, να υιοθετήσει νομοθετήματα και με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπρόσωποι των, της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες να μπορέσουν να ξαναπάνε στη Λιβύη και να εργαστούν εκεί και να ληφθεί υπόψη και να αρχίσει να λειτουργεί η Συμφωνία Επιστροφής ε, και αυτό θα σήμαινε ότι το Συμβούλιο φαίνεται ότι έχει εγκαταλείψει τέτοιου είδους ε, αιτήματα σε μια χώρα συγκεκριμένα όπου καταπατούνται κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα καθημερινά. Η Ιταλική αυτή εξαίρεση δεν μπορεί να γίνει ο κανόνας για τα, τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι λίγο αξιόπιστο να συνεχίσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμικοί φορεί να θέλουν να συνάψουν με συμφωνία πλαίσιο με δικτατορική χώρα όπω η Λιβύη. Δεν μπορούμε να ξεκολουθούμε να λέμε ότι η Λιβύη έχει εμπορικέ σημαντικέ σχέσει με τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και διαδραματίζει ρόλο εταίρου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω όσον αφορά τη λεκάνη τη Μεσογείου και να θέσουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σαν δευτερεύουσα σημασία. Η πρώτη προπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει αξιόπιστο διάλογο με τη Λιβύη είναι να επικυρωθεί η Σύμβαση τη Γενέβη από αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε να, βάζουμε, να ανταλλάσσουμε τα οικονομικά συμφέροντα με τι ανθρώπινε ζωέ, όχι μόνο των πολιτών τη Λιβύη, αλλά και των πολιτών που ξεφεύγουν από άλλε χώρε και διότι ξεφεύγουν από τη σκεφτική δίωξη και διώξει και αντί να βγουν καταφύγιο στη Λιβύη βρίσκουν βασανιστήρια και θάνατο. Δεν πρέπει να λησμονούμε τι χιλιάδε τίματα βοήθεια που ζητούν ε, οι κρατούμενοι στι φυλακέ τη Λιβύη. Να λησμονήσουμε τη φρίκη ε, των φυλακών του Καφούκη που όταν πήγαμε εκεί ε, δεν έχουν πολλά πολιτικά δικαιώματα όπω ελευθερία έκφραση, ε, του συνεταιρίζεστε οι, οι πολίτε τη Λιβύη. Η, η προφορική τροπολογία τη αιτιολογική σκέψη Β θα πρέπει ε, ε, ναι, λοιπόν, ε, είναι κάτι που δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε λοιπόν το πρότυπο τη Ιταλική Συμφωνία. Εμεί θα το καταψηφίσουμε. Συμφωνία Ιταλία και Λιβύη είναι πολύ πιο περίπλοκη συμφωνία με σαφεί προποθέσει που αφορούν θέματα πολύ πιο περίπλοκα από την κοινή ε, περιπολία των ακτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξακολουθήσει να είναι αξιόπιστο πρέπει να λέει τα πράγματα με τα ονόματα του, παρόλο που αυτό μπορεί να είναι ενοχλητικό. Λοιπόν, θα πρέπει η πατριαρμοστία τη πρόσφυγε να μπορεί να παίξει ελεύθερα το ρόλο στην περιοχή και θα πρέπει το τη Λιβύη ε, να, να του αφήσει να κινηθούν. Επ' αυτή τη βάση δάσο που θα μπορούμε να συνάψουμε συμφωνίε. Δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε ούτε με του δικτάτορε ούτε με του τρομοκράτε. Είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι το Συμβούλιο ε, τη Διοίκηση, ε, του Διοικητικού Συμβουλίου ενό κολοσσού οικονομικού, μια εταιρεία οικονομική. Να ευχαριστήσω την κυρία Γκομέζ. Μας δίνει ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις που είναι κάπως ε, ε, αστείες γιατί ε, ε, μας επισημαίνεται από τα όσα γίνεται στην την Ισία ότι δεν είναι δυνατόν έτσι εύκολα να εκφράζουμε ικανοποίηση και να θεωρούμε ότι ένα τέτοιο καθεστώς είναι αποδεκτό και να τολμούμε να σχεστίζουμε με ένα τέτοιο καθεστώς το χαρακτηρισμό σεβασμό των δικαιωμάτων γιατί δεν σέβονται τίποτα. Εγώ λέω και περισσότερες ακτές μας και όλοι Όλοι μας λένε με τον ένα τον άλλο τρόπο ότι καλύτερα να πνιγούν παρά να γυρίσουν πίσω γιατί υπάρχει προβασανιστήρια, βιασμοί, επαναπροωθήσει, ρατσισμό, ρατσισμός, όλα, όλα αυτά. Αυτός ο, ο κατάλογος των φρικτών πραγμάτων που υφίστανται οι μετανάστες στη Λιβύη. Αλλά δούμε τι να κάνουμε, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ε, επιτακτικό, αφορά και την υποτιαρμοστία να καλυφθούν όλοι αυτοί τους οποίους ε, λέω ότι πρέπει να καλυφθούν η υπατιαρμοστία ε, όλοι αυτοί οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθειά μας να τη δώσουμε τώρα όσον αφορά την νομιμοποίηση όλων αυτών που μπαίνουν στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος γιατί πρέπει να δούμε πρώτα πρώτα ποιοι είναι οι στόχοι που επιτάσσει η συνθήκη ότι πρέπει να διέπουν την εξωτερική μας πολιτική. Κάμπελ. Το 2007 πρόεδρε. Που δεν σαρκωσεί. Λοιπόν δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της απελευθερίας των πέντε νοσοκόμων και της ε, πόλης εκείνων των πυράβλων για εκατοντάδες εκατομμύρια. Είχαμε και τη βόμβα στο αεροπλάνο που έφυγε στο Λόκερμπι και είχαμε και το γιο του Καντάφη που είπε ότι ε, τελικά η αγορά των όπλων έγινε αντί των της των φυλακισμένων. Ήταν deal. Οι Times λένε ότι η κυρία Άστον θέλει να σταματήσει να υπάρχει το εμπάργο που ξεκίνησε με την Κινάν Μέν και λέει ότι λέει η κυρία Άστον ότι αυτό εμποδίζει την περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι εμπόδιο στο να σωθεί το ευρώ. Και αντιστοίχω και για τη Λιβύη θέλει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει το Euro γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά των Κινέζων για να το σώσουν που τώρα χαλαρώνει ε, η επιτήρηση όσον αφορά τη Λιβύη και έχουμε αυτά τα 2,9 εκατομμύρια. Ε, τα οποία δόθηκαν για πορτογαλικά, ισπανικά και ελληνικά ομόλογα. Όμως σε αυτές τις χώρες εκτελούνται εκατομμύρια. Κάθε μέρα τόσο κόσμος, ειλικρινά πέστε μου, πόσο χαμηλά θα κατρακυλήσει η Ευρωπαϊκή για να σώσει το ευρώ. Ο κύριος Μέλτσερ για ένα λεπτό. Κύριος Μέλτσερ, ευχαριστώ πρόεδρε. Η εξέγερση στην Τινησία συγκλώνησε και τις γειτονικέ χώρες του Μαγκρέπ και τη Λιβύη χώρες που είναι δικτατορικά καθεστώτα. Σίγουρα μια τέτοια ανατροπή είναι μια ευκαιρία για το δημοκρατικό καθεστώς, για τη δημοκρατία. Ωστόσο μόνο τότε αν δεν την εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία οι Ισλαμιστές. Σίγουρα αυτά θα έχουν και επιπτώσεις ε, στις ε, ε, ροές των προσφύγων. Μια συνεργασία των Αφρικανικών χωρών όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι σημαντική υπόθεση και για την Ένωση και την βοήθεια των κρατών αυτών για την αντιμετώπιση της παραγωγής παράνομης μετανάστευσης ε, πρέπει να πούμε ότι ακολουθείται η λαθασμένη πορεία. Και έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυξιακή βοήθεια και αυτή η αναπτυξιακή βοήθεια το πλαίσιο της πρέπει να επανεξεταστεί για να μην υποφελούνται δικτατορικά καθεστώτα και τα διεφθαρμένα καθεστώτα αλλά να υποφελούνται οι πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει σε σχέση με την αρνητική αυτή κατάσταση που επικρατεί στις ε, χώρες του αραβικού κόσμου να δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Vorsitzender. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Έχουμε ευθύνη έναντι όλων των γυναικών, των παιδιών, των ανδρών που ζητούν προστασία λόγω τη κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Αυτή η ευθύνη απορρέει αφενό λόγω ηθικών αξιών, επί των οποίων οικοδομείται και βασίζεται η Ευρώπη, και λόγω και τη ιστορία μα, που πολύ συχνά την ξεχνάμε εμεί οι Ευρωπαίοι. Και από την άλλη πλευρά και λόγω εγγυήσεων, λόγω διεθνών συνθήκων. Όποιος έχει ευθύνες πρέπει να είναι πρόθυμος να υπομειστεί και το βάρος αυτών των ευθυνών. Αυτό σημαίνει ε, προθυμία των κρατών μελών να συμμετάσχουν και στην οικονομική προσπάθεια. Δεν είναι δυνατόν όμως ε, να φορτώνονται όλα στις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τέτοιου είδους καθεστώτα να πληρώνονται όπως το καθεστώς του Γκαντάφη ώστε να προλαμβάνουμε αυτή την επιβάρυνση, αυτό το άχθος προσφύγων ε, και μεταναστών στην Ευρώπη. Εδώ ρισκάνουν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι. Όμως αυτό το καθεστώς δεν ενδιαφέρεται για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι ή να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Πρόκειται για ψυχρό υπολογισμό οικονομικού κέρδους. Και εδώ θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι καταπιέζονται, καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα κατάφορα. Είχα πάει εγώ σε καταβλισμούς και στρατόπεδα σε σχέση με πρόσφυγες και μετανάστες. Δεν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα όμως εκεί. Μας λένε δεν παίρνουν ε, ε, κανονιοφόρους ε, για ε, να προστατεύουν καλύτερα τα σύνορά τους ε, και πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Και τώρα επειδή έχουμε οικονομικά ωφέλη ή υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας επανεισδοχής προδίδουμε τις αξίες μας. Αυτό είναι απαράδεκτο και πιστεύω ότι αυτή η εντολή για τις διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι προσπελάσιμη, να είναι στη διάθεση όλων των Ευρωβουλευτών και όχι μόνο στη διάθεση κάποιων. Δεν μπορεί να υπάρχει μυστική διπλωματία. Είναι απαράδεκτο να έχουμε τέτοιου είδου σχέσεις με ένα καθεστώς, καθεστώς του Καντάφη. Και αυτό είναι ένα σημείο που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και ζητώ από εσάς και η Άννα Γκόμε ανέφερε όλα τα στοιχεία και τα σημεία που πρέπει να είναι σεβαστά προηγούμενα προτού καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τον Καντάφη. Ευχαριστώ. Έχουμε τρεις ομιλητές. Ο πρώτος είναι ο ε, Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εκείνοι που είναι κατά μια συμφωνία με τη Λιβύη πρέπει να καταλάβουν ότι είναι γειτονέ μας και δεν μπορούμε να γνωρούμε τους γειτονέ μας, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να συμβιώνουμε. Ακόμα και αν δεν μα αρέσουν τα πάντα για αυτούς και τα όσα κάνουν. Είναι πολύ εύκολο εκείνοι οι συνάδελφοι που δεν προέρχονται από χώρε που είναι γείτονε τη Λιβύη να μιλούν κατά αυτή της συμφωνία. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για εκείνους που ζουν σε χώρες της Μεσογείου που είναι κοντά στη Λιβύη γείτονές τους και πρέπει να βρουν τρόπο να συνεργαστούν με αυτή τη χώρα. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και ένα κεφάλαιο περί μεταναστεύσεως και μια συμφωνία για την επανεισδοχή. Ταυτόχρονα ε, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα για διεθνή προστασία εκείνων που ετούν άσυλο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίλαν Μον για ένα λεπτό. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση για την Λιβύη λαμβάνει χώρα να έχουμε πάρα πολύ σημαντικέ αλλαγέ που γίνονται σε άλλη γειτονική χώρα, την Τινησία. Ε, Ανέκαθεν ναι, θεωρούσαμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθά να έχουμε τέτοιε μεταρρυθμίσει στην Μεσόγειο. Και ο στόχο είναι να υπάρχει χώρο ευημερία και ελεύθερα και σα παραπέμπω στα όσα έχω πει όλα αυτά τα χρόνια και επαναλαμβανημένα έχω πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυνατόν να προσανατολίζεται μόνο προς μονοδιάστατη πολιτική χρειάζεται μόνο να γίνει αυτή η συμφωνία πλαίσιο να συνεργαστούμε ανθρώπου με μεταναστευτικές ροέ και να γίνει και επίση και συμφωνία επανεισδοχή των λαθρομεταναστών να καλύψουμε και του ε, ηθογενεί τρίτων χωρών ακριβώ όπω γίνεται σε όλε τι συμφωνίε επανεισδοχή να υποχωρήσουμε σε αντίθετη γνώμη που έχουν οι Λίβοι θα ήταν πάρα πολύ κακό ε, δεν θα θεωρούσαμε ότι είναι χώρα μετάβασης και θα ήταν προηγούμενο κακό για Αλγερία και Μαρόκο συμφωνία τον οποίο η πορεία έχει κολλήσει εδώ και χρόνια άρα θα πρέπει να επιμείνουμε προς τους Λίβιους να σεβαστούν τα δικαιώματα των, ε, των προσφύγων και επίσης την αρχή της μη επαναπρόθεσης. Τέλος ο κύριος Γιακολίνο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στο Μαγκρέμπ περνάνε μια πολύ δύσκολη φάση. Συγκρούσει σε ματηρέ των τελευταίων ημερών στην Τινησία είναι η απόδειξη αυτή, η κραυγαλαία. Θα ήταν πάρα πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή την ιστορική να μην λάβουμε υπόψη τις απαιτήσει, τις ανάγκες, τις μεγάλες για την ενίσχυση των σχέσεων με τη Λιβύη που είναι στη Μεσόγειο και έχει ένα θεμελιώδη ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά τη συγκράτηση και τη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών με όλε τι αντιθέσει που υπάρχουν εκεί. Εγώ είμαι στη Λιβύη με τη συνάδελφο Γκόμε και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια συμφωνία πλαίσιο θα μπορούσε σίγουρα να συμβάλλει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην εφαρμογή θεμελιωδών ελευθεριών και στο θέμα το ενεργειακό. Το να μην προστραφούμε προς το Μαγκρέπ και τη Λιβύη θα ήταν κάτι που θα ήταν σοβαρότατο σφάλμα. Ένα πρότυπο αναφοράς είναι η συνθήκη φιλία τη στο Ιταλικό που θα μπορούσε να εφαρμοστεί για να εγγυηθεί συγκεκριμένα ότι θα εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο, το, η συμφωνία πλαίσιο. Εξ ονόματο της Επιτροπής, ο κύριος Φούλη έχει το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα σχόλιά τους και θα ήθελα επίσης να πω προς την εισηγήτρια την κυρία Γκόμες ότι θα της στείλω περισσότερες λεπτομέρειες για τα διάφορα εθνικά ενδεικτικά σχέδια για το 2011 μέχρι 2013 που προβλέπουν 60 εκατομμύρια ευρώ που θα χορηγηθούν από τα προγράμματά μας για τη Λιβύη. Έχω πλήρη επίγνωση ότι κάποια θέματα είναι προβληματικά όσον αφορά τις σχέσεις με τη Λιβύη. Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε τη δημιουργία σχέσεων με τη Λιβύη για να μπορέσει να συζητήσει όλα τα θέματα ανοιχτά και επικοδομητικά και τα πιο ευαίσθητα ακόμα συμπεριληφθούν, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός θεμελιωδών ελευθεριών, όλα τα δικαιώματα των μεταναστών. Επεσκέφθην με τη Σεσίλια Μάλστρομ το κέντρο κράτησης στη Λιβική έρημο πέρσι. Οπότε δεν τρέφω αυταπάτες. Καμία αυταπάτη όσον αφορά τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είχα τη δυνατότητα επίσης να κατανοήσω τις αναλλακτικές λύσεις αλλά έχουμε ξανά την μετανάστευση. Να πω τώρα κάτι, ένα τρίτο προσωπικό σχόλιο να αναφέρω. Στις διαπραγματεύσεις ε, προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και τις αξίες μας, αυτές τις οποίες πιστεύουμε. Ε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η Λιβύα έδειξε την προθυμία να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούμε αυτό ότι είναι κάτι θετικό και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να ακολουθεί αυτή την πολιτική των συνομιλιών. Βεβαίω, εγώ είμαι δεσμευμένος ότι να εξασφαλίσω ότι όλα αυτά θα γίνουν με διαφάνεια, λαμβάνοντα υπόψη τι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Finally, taking the και τέλος, αναλαμβάνοντας την ε, Προεδρία, έχω να ζητήσω τώρα από την εισηγήτρια Άννα να συνοψίσει τα της ε, εκθεσιώς της. Ε, εγώ ευχαριστώ όλους που έλαβαν μέρος. Φάνηκαν όλα μας τα διλήμματα από τη συζήτηση, αλλά πρέπει να σας πω ότι έμαθα όταν πήγα στη χώρα με την αντιπροσωπεία μας, με επικεφαλής τον φίλο Παντζέρετ, πριν από λίγους μήνες ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την ρότα που έχουμε δεσμευθεί και να αναγνωριστούν οι δυσκολίες για το πόσο δύστροποι είναι οι συνομιλητές μας. Έχουμε ανθρωπιστική υποχρέωση προς τον λαό της χόλας που τόσο υποφέρει. Και ιδίως οι μετανάστε αυτοί που θέλουν να περάσουν μέσα από τη χώρα και υφίστανται αυτά που υφίστανται μεγάλες δυσκολίες και δυσκολίες υφίστανται στο ότι αυτοί το καθεστώς ήταν σε κατάσταση απομόνωσης όλες οι προϋποθέσεις και όλοι που τάσουμε θα πρέπει να, μην πάψουν να συνεχίσουμε την ίδια ρότα και γι' αυτό σας λέω. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί έτσι αυτή η αντιπροσωπεία. Όπως είπαν πολλοί από εσά. αυτό το οποίο είναι στην Τινησία θα έχει επιπτώσεις και στην Λιβύη παρά τις διαφορές γιατί βέβαια υπάρχουν διαφορές αρκετές γιατί εξαρτώνται τελείως στην Λιβύη από το πετρέλαιο. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές οπτικές γωνίες, όμως θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την πορεία των αποτεύξεων από την Κομισιόν. Ευχαριστώ για το όσα είπατε, την χρήσιμα από την Επιτροπή. Θα προσπαθήσουμε να κατεβάσουμε προτάσεις προς εσάς και θα πρέπει να δούμε πώς θα πετύχουμε μια ευρεία συνένεση. Θα συνεργαστώ και με τους σκιώδεις εισηγητές Άρα θα πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα προς Κομισιόν Συμβούλιο και προς τους Λιβύους συνομιλητάς για όλα τα θέματα που θεωρούμε σημαντικά και όπου θέλουμε να επιτευχθούν βελτιώσεις και στις διμερείς σχέσεις αλλά και στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Αυτό είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ευρωβουλευτά και ευχαριστώ επίσης και για όλες τις παρεμβάσεις. Και έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το σημείο στη συζήτηση. Αύριο στις 12 η ώρα θα διεξαχθεί